I think we can start. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίζω θερμά στη σημερινή μας σε την Επίτροπο για θέματα μεταφορές, την κυρία Μπούρτς, η οποία θα μας παρουσιάσει σήμερα το πακέτο για τις ενέργειες μεταφορές που έχει θετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι καλό το γεγονός ότι επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει την δραστηριότητα και την πρωτοβουλία σε αυτό το θέμα των ενέργειων μεταφορών. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις και να ε, δώσουμε λύσεις στα προβλήματα για τις ενέργειες μεταφορές, παραδείγματι αυτά που προκύπτουν από την όλο και ενισχυόμενη διάδοση των μη επανατολμένων τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων, ενέργειων οχημάτων. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την αηφορία των ενέργειων μεταφορών. Πρέπει να φροντίσουμε η ευρωπαϊκή αεροβιομηχανία να ε, καταστεί ανθεκτική στη διεθνή, ε, στον διεθνή ανταγωνισμό. Και γι' αυτό, για να μας δώσει τις απαντήσεις ε, η κυρία Επίτροπος, την έχουμε προσκαλέσει, θέλω να επισημάνω ότι ορίζεται από τη συνθήκη Λισαβόνα στο άρθρο 218 ότι συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό θέλουμε να έχουμε έγκαιρη συμμετοχή στη διαδικασία, όχι εκ των υστέρων, όχι όταν πια είναι πολύ αργά και να είμαστε σε θέση να πούμε ε, ότι κάτι μας βρίσκει σύμφωνος ή όχι από τις λύσεις που έχετε να προτείνετε. Δηλαδή να μην συμβεί αυτό που συμβαίνει με το TTIP. Κυρία Μπούρτ, σας ευχαριστώ και πάλι που είστε εδώ και για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία. Περιμένουμε με αδημονία την παρουσία σας. Παρακαλώ. Thank you very much, uh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κράμερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα με σκοπό να συζητήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό πακέτο το οποίο θα δρομολογήσουμε σήμερα και πρέπει να πω ότι πραγματικά πρώτα το παρουσιάζω σε εσά και μετά στο Συμβούλιο. Αλλά μετά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ξέρω όμω ότι ήδη γνωρίζετε κάθε αράδα. Είχατε την ευκαιρία να το μελετήσετε. Σοβαρά τώρα, το πακέτο αυτό είναι για μας πολύ σημαντικό. Θα το επαναλάβω, είμαι περήφανη και πολύ ευτυχής που καταφέραμε να το περάσουμε και είμαι περήφανη γιατί είναι το αποτέλεσμα μιας ε, συμμετοχής ε, όλων και δέσμευσης όλων των εμπλεκομένων φορέων, του τομέα των ε, οικοσυστημάτων, ε, της αεροπορίας ε, και οποιοδήποτε συμμετέχει στο πλαίσιο αυτό και στον κλάδο αυτό, συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί όντως υπήρχαν προβλήματα. Χαίρομαι επίσης επειδή υπάρχει και ένα σχέδιο δράσης που συνοδεύει το έγγραφο αυτό επί τη βάση όλων αυτών θα ήθελα να σας πω ότι θα είμαστε, πιστεύω, πολύ παραγωγικοί στο μέλλον. Να πω ορισμένα αριθμητικά στοιχεία θα ήθελα να σας παραθέσω, γιατί είναι σημαντικά για να μπορέσετε να καταλάβετε το πεδίο εφαρμογής αυτής της στρατηγικής για την αεροπορία, να καταλάβετε όλα τα στοιχεία που το συνθέτουν. Πρώτον, Δύο εκατομμύρια άνθρωποι στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολούνται στον τομέα αυτών και πιστεύουμε ότι υπάρχει δυναμικό για πολύ περισσότερους. Παράλληλα όμως υπάρχει και ένας κίνδυνος ε, αν δεν συνεχίσουμε ε, την εξέλιξή μας και την ανάπτυξή μας υπάρχει περίπτωση να, υπάρξει να υπάρξουν πολλές αρνητικές συνέπειες. Κάτι ακόμη, άλλο στοιχείο σημαντικό είναι ότι πάνω από 110 δις ε, ε, ε, σε, ΑΕΠ εκπροσωπεί η αεροπορία. Θέλουμε βέβαια πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή της αεροπορίας στο ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα. Είναι πάντως ήδη μεγάλο το ποσό. Τρίτον, η αεροπορία είναι το μοναδικό μέσο μεταφοράς κατά πολύ ε, που επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες ε, να ε, μπορούν να μετακινούνται από πολύ απομακρυσμένες περιοχές, δηλαδή για αυτούς είναι ο μοναδικός τρόπος μεταφοράς και ειδικότερα για τον τομέα του τουρισμού πρέπει να πω ότι υπάρχει μια, είναι μια πολύ σημαντική συνιστόσα γιατί για αυτούς τους ανθρώπους η αεροπορία δημιουργεί δουλειά θέσεις αποσχόλησης και φυσικά μπορεί να ε, δημιουργήσει και ε, περισσότερα έσοδα στις πολύ απομακρυσμένες περιοχές. Πάνω από 510 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό που επιφέρει ε, η αεροπορία στον τουρισμό. Ελπίζουμε ότι θα εξακολουθήσει να ισχύει αυτό και ότι θα υπάρξουν οι συνθήκες που θα επιτρέψει ε, που θα, θα υπάρξουν συνθήκες που θα επιτρέψουν σε αυτόν τον κλάδο της ευρωπαϊκής οικονομίας να αναπτυχθεί περαιτέρω. Εκτός ε, από τα στοιχεία που αφορούν ε, τα περιβαλλοντικά και το οικοσύστημα, ελπίζουμε ότι θα υπάρξει και επίπεδο υψηλότερο ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκή αεροπορίας σε παγκόσμιο επίπεδο γιατί αυτό είναι μια τεράστια ευκαιρία όχι μόνο για τους ε, υπάρχοντες ευρωπαϊκούς παίκτες, αλλά είναι μια τεράστια ευκαιρία και για μελλοντική εξέλιξη. Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο λοιπόν υπησέρχεται η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με εσάς. Και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας θα ήθελα να σας πω ότι, να σας ευχαριστήσω μάλλον ότι ήσασταν πάρα πολύ επικοδομητικοί ήταν ε, κρίσιμη και επικοδομητική η συνεργασία σας και ελπίζουμε ότι σε αυτό το πνεύμα θα παραμείνει η συνεργασία μας και για το μέλλον. Χαίρομαι με το ψήφισμα για τη στρατηγική της αεροπορίας το οποίο υπερψηφίσατε με συντριπτική πλειοψηφία στις 11 Νοεμβρίου. Για μένα αυτό ήταν μια πολύ σημαντική όθηση και μου έδειξε ότι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, ότι έχουμε ε, σκοπό να επιτύχουμε τους ίδιους, τους ίδιους στόχους και ελπίζω ότι η συνεργασία μας θα μας επιτρέψει στο μέλλον ε, να ε, περάσουμε και στην πραγματική λειτουργία όλων αυτών των στοιχείων της στρατηγικής. Για ποιο λόγο υποβάλλουμε αυτό το περιεκτικό πακέτο. Είχαμε υπόψη μα πέντε προτεραιότητε Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και αναρωτιόμασταν συνεχώ τι υποστηρίζουμε. Ανάπτυξη και θέσει απασχόληση, επενδύσει, να προσελκύσουμε επενδύσει στην Ευρώπη. την περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανικής μας υποδομής που τη χρειάζεται οπωσδήποτε η Ευρώπη. Υποστηρίζουμε την ε, περαιτέρω ε, προώθηση της ε, ενιαίας αγοράς που είναι βασική συνιστόσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, υποστηρίζουμε περαιτέρω την Ενεργειακή Ένωση και την κλιματική αλλαγή και τις σχετικές υποχρεώσεις. Και πρέπει να σας πω ότι πραγματικά χαίρομαι για τον τρόπο με τον οποίο μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στις ε, πέντε αυτές προκλήσεις. Θα ήθελα καταρχάς ε, να αναφερθώ στην Ευρώπη ως παγκόσμια δύναμη. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί, Γιατί η ανάπτυξη στον τομέα της αεροπορίας κατά τα ερχόμενα έτη θα είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασία, Λατινική Αμερική, Τουρκία, τις χώρες του Περσικού κόλπου και ενδεχομένως ε, στην Αφρική ε, σε ένα πιο μακροπρόθεσμο ε, μέλλον. Η Ευρώπη επίσης αναμένεται να σημειώσει ανάπτυξη, αλλά επειδή είμαστε πολύ όρημη αγορά, η ανάπτυξη στην Ευρώπη θα είναι μικρότερη από ό,τι σε, άλλες, σε άλλα μέρη του κόσμου. Γι' αυτό το λόγο σε επίπεδο διεθνών δραστηριοτήτων αυτό που θα θέλαμε να προωθήσουμε είναι περιεκτικές συμφωνίες με τις χώρες με τις οποίες θέλουμε καλύτερη ε, διασύνδεση και αναφέρομαι στην Ασία, τις χώρες ΑΣΕΑΝ και την Κίνα. Αυτές είναι οι χώρες που είναι στον κατάλογό μας. Έχουμε σκοπό να προτείνουμε περιεκτικές συμφωνίες με τις χώρες αυτές. Επίσης, χώρες του Περσικού κόλπου, Μεξικό, Βραζιλία και στην Ευρώπη οι δύο κυριότεροι εταίροι είναι η Τουρκία και η Γερμανία. Με αυτούς, με αυτές τις δύο χώρες ε, θα επιδιώξουμε συμφωνίες περιεκτικές. Θα ζητήσουμε από το Συμβούλιο να μας βοηθήσει, να μας υποστηρίξει και να μας δώσει μια δυναμική εντολή βάσει της οποίας μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Μια περιεκτική συμφωνία, όπως είπα, που θα μας επιτρέψει να αναπτυχθούμε, αλλά να αναπτυχθούμε υπό τις συνθήκες για να δούμε, να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και τα αποτελέσματα ε, μεσοπρόθεσμα στο μέλλον. Υπάρχει ανάγκη ενός ρυθμιστικού πλαισίου, ενός ρυθμιστικού περιβάλλοντος και Βεβαίω, θεωρούμε ότι οι περιεκτικές συμφωνίε είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, γιατί θα μας δώσει τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε τα βασικότερα σημεία για να εξασφαλίσουμε δύο βασικά στοιχεία, την αμοιβαιότητα και το ισότιμο πεδίο. Αυτό ε, για μας, ε, αυτά τα δύο στοιχεία είναι βασικά στοιχεία ε, των συμφωνιών αυτών εκτός από τη σχέση της ε, ευρωπαϊκής αεροπορίας ε, σε διεθνές επίπεδο, το δεύτερο στοιχείο είναι η ενιαία αγορά. Εκεί προσπαθήσαμε πάρα πολύ να εξαλείψουμε τα εμπόδια για έναν ακόμη ισχυρότερο ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, για πραγματική ενιαία αγορά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βασικό στοιχείο το οποίο μας απασχολεί είναι η συμφόρηση και στο έδαφος αλλά και στον αέρα. Γνωρίζουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος δεν είναι ο χώρος ε, που την χάνει της αποτελεσματικότερης ε, χρήσης και αξιοποίησης και ελπίζουμε να ε, συνεργαστούμε με εσάς, να προσπαθήσουμε να λύσουμε κάποια θέματα ας πούμε νομοθεσίας που δεν εφαρμόζεται σωστά ή δεν εφαρμόζεται καθόλου για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικές πτήσεις, όχι πτήσεις ε, zigzag, αλλά πτήσεις τις οποίες μπορούμε πραγματικά να τις διαχειριστούμε καλύτερα, να διαχειριστούμε και τους αερολιμένες καλύτερα, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη θα προκύψει και από καλύτερη διαχείριση, όχι μόνο από επιπλέον υποδομή. Τώρα, το κόστος του καταχειρματισμού. Σας το λέω για να σας εξηγήσω για ποιο λόγο έχουμε τόσο ισχυρή άποψη για το θέμα αυτό. 5 δισεκατομμύρια κατ' έτος. Έχουμε την πολυτέλεια, είμαστε τόσο πλούσιοι ώστε να μπορούμε να πετάμε, να σπαταλάμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Απλώς και μόνο γιατί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, δεν μπορούμε να βρούμε μια κοινή λύση. Ελπίζω ότι αυτό θα αποτελέσει κίνητρο για μας και ότι θα κάνουμε πολύ πιο αποφασιστικά βήματα προς την κατεύθυνση της εφαρμογής των απαραίτητων δράσεων. Κάτι ακόμη που θα ήθελα να σχολιάσω. Το κόστος της αδράνειας είναι 880.000 θέσεις εργασίας ε, που θα χαθούν. Δεν θέλω να φοβήσω κανέναν, αλλά αν δεν προχωρήσουμε, αντί να πάμε προς τα θα υπαναχωρήσουμε. 52 δις ευρώ μέχρι το 2035 χαμένου ΑΕΠ. Ελπίζω ότι αυτά τα στοιχεία να είναι αρκετά για να αποτελέσουν κίνητρο για μας. Οπότε κάνω έκκληση και σε εσά και στο Συμβούλιο να εγκρίνετε τον αναθεωρημένο κανονισμό για τις ε, χρονοφυρίδες για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα για κτήσεις και για να μπορέσουμε να έχουμε έναν αποτελεσματικό εναέριο χώρο. Έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο στοιχεία ήδη μπροστά μας και πρέπει να δούμε σε επιχειρησιακό επίπεδο πώς θα τα προωθήσουμε. Πρέπει να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλες μας τις ευκαιρίες στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, γιατί αυτό θα μας καταστήσει ισχυρότερους όταν πρέπει να ανταγωνιστούμε και ενδεχομένως να ηγηθούμε της παγκόσμιας αεροπορίας. Πέντε τομείς ε, που αναφέρονται και στη στρατηγική πιστεύω ότι χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και αναφέρονται στην εσωτερική μας αγορά. Πρώτον, τα δικαιώματα των επιβατών. Πρέπει να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό. Δεύτερον, περιβαλλοντικός αντίκτυπος. Προσπαθούμε να το προωθήσουμε μέσω του ΙΚΑΟ. Το 2016 είναι πάρα πολύ σημαντικό έτος γιατί θα γίνουν πολύ σημαντικές διαπραγματεύσεις οι οποίες θα καθορίσουν τη σχέση μας σε παγκόσμιο επίπεδο με, τις, με τους υπόλοιπους εταίρους. Τρίτον, περισσότερα προδιαγραφές για ασφάλεια, για ασφάλεια από κακόβουλες πράξεις, και επίσης το άνοιγμα της αγοράς πρέπει να μην ξεχνάμε κάθε φορά που ανοίγουμε την αγορά μας, να μην ξεχνάμε τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά στοιχεία. Τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να λειτουργήσουν. Και γι' αυτό χαίρομαι όλος ιδιαιτέρως που όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφωνούν μαζί μας και θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας για να βρούμε καινούριου τρόπους να προχωρήσουμε. Η στρατηγική μας λοιπόν προτείνει σημαντικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, αναβάθμιση των ευρωπαϊκών κανόνων ασφάλειας, ώστε να υπάρξουν προδιαγραφές ε, ασφάλειας υψηλότερες όσο αυξάνεται και ο όγκος της κυκλοφορίας, χρειάζεται ένα αποτελεσματικό, αποδοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο που θα δώσει τη δυνατότητα στην αεροπορία να ε, είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά να αντανακλά και τον κοινωνικό διάλογο, τον οποίο εμείς ε, θεωρούμε ότι βρίσκεται στον, στο επίκεντρο όλων των συζητήσεών μας. Γνωρίζω ότι όλα αυτά τα ζητήματα είναι πολύ σημαντικά για εσάς και προσβλέπω στη συνεργασία που θα έχουμε, ώστε να έχουμε και μια ταχεία εφαρμογή, υλοποίηση από του χρόνου. Τη στρατηγική. Το τέταρτο σημαντικό στοιχείο. Πέρα από τη διεθνή την εσωτερική αγορά για τα πρότυπα, είναι η καινοτομία. Σήμερα η καινοτοπία είναι κινητήριος μοχλός της ε, διεθνούς οικονομίας, όχι μονογραμμικά αλλά και ως προς τη βιωσιμότητα. και η καινοτομία μαζί με την ψηφιοποίηση που είναι βασικό της συστατικό είναι κεντρικά στοιχεία που επιτρέπουν κεντρικοί enablers αυτής της στρατηγικής και της υλοποίησής της. Χρειάζεται λοιπόν η άσα να ενέχεται νωρίς από την αρχή την ώρα διαδικασίας και αυτό θα είναι μια βασική ωφέλεια για τις επιχειρήσεις. ο χρόνος που έχει κανείς για να παραδώσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του και να επικαιροποιήσει τις ε, παραγωγικές του διαδικασίες είναι κρίσιμος. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που είναι αναβιώμενες νέες τεχνολογίες και η χρησιμοποίηση των drones που στοιχειοθετούν, αν θέλετε, μια πλατφόρμα εντό τη οποία θα πρέπει να κινηθούμε στα πλαίσια δηλαδή τη στρατηγική αυτή για την αεροπλοεία. Αλλά στο πλαίσιο αυτό πάνω απ' όλα προσπαθούσαμε να επιτύχουμε μια ισορροπία μεταξύ ασφάλειας αφενός, ασφάλειας δικαίου αφετέρου και προστασίας των πολιτών και των δεδομένων. Όλα αυτά είναι τμήμα της επανεξέτασης ε, του βασικού κανονισμού ΕΑΣΑ και καθότι μου είπαν ότι ήδη έχω μακρηγορήσει, δύο ακόμα στοιχεία θέλω να αναφέρω που είναι πολύ σημαντικά. Οι επενδύσεις γιατί οι αερομεταφορείς και οι κατασκευαστές Ελπίζουμε ότι θα είναι πιο εύκολο για αυτούς μέσω της ε, στρατηγική αυτή να έχουν πρόσβαση σε νέες αγορές. Και θεωρούμε ότι οι ε, ολοκληρωμένε συμφωνίε θα είναι ένα πολύ καλό μέσο ή στο πλαίσιο αυτό. Και για τον 2008 μέχρι 2008 θα έχουμε επικαιροποίηση των διατάξεων των κανονισμών ώστε να επιφέρει καλύτερη, πληρέστερη ασφάλεια δικαίου για όλους τους ε, επαγγελματίες. Έχουμε και τον 868 για την αντιμετώπιση των στρεβλωτικών ή άνισων πρακτικών στην αγορά και αυτό που σκοπεύουμε να το κάνουμε μέχρι το 2016. Μετά έχουμε τις θέσεις απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 30 εκατομμύρια ευρώ ανά μέχρι το 2020 σκοπεύει να επενδύσει εδώ. Και όχι μόνο ως εργαλείο διαχείρισης αν θέλετε της κυκλοφορίας, αλλά ως ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα εξαγωγής. Και ελπίζουμε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία 300 και άνω χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας αλλά κυρίως και να συμβάλλει και στην, ε, στον περιορισμό, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επομένως, για να κλείσω, θα πω ότι η στατική αυτή σχεδιάστηκε και καταρτίστηκε ώστε να ενέχει ωφέλειες για όλους τους, για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, για τους πολίτες, καλύτερη ασφάλεια, καλύτερες τιμές κόστος πτήσεων, καλύτερες συνδέσεις στις πτήσεις. Και από την ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να στοχεύσουμε στην διεθνή αγορά ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τους εθέρες του κόσμου και για τις αεροδρομικές αεροπορικές συνδέσεις με συγχωρείτε ώστε να βασίσουμε την προσέγγισή μας υπό την έννοια της ασφάλειας ε, σε μια βασική σχέση κόστους ωφέλους. Πρέπει να ενισχύσουμε επίσης τον κοινωνικό διάλογο της πολιτικής αεροπλοείας και να λάβουμε υπόψη μας όλες τις καλές ιδέες που θα προκύψουν από το διάλογο αυτό. Και χρειαζόμαστε όλους τους, αερο... τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχουν ενεργά στο διάλογο αυτό και να ενισχύσουμε και την απασχόληση στον τομέα μέσω της καινοτομίας. Δημιουργούμε δυνατότητες θέσεων απασχόλησης υψηλή αξίας. Θέλουμε επίσης μια, ένα σαφές και ασφαλές πλαίσιο δικαίου και για τους αερομοτεφορείς νέες αγορές μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και το European Sky είναι πραγματικά μια χρυσή ευκαιρία να διαχειριστούμε καλύτερα τον οικονομικό αντίκτυπο της δραστηριότητας αυτής. Και ο διαφρομένος διάλογος που ήδη είχαμε μαζί τους μας έχει δώσει συμπληρωματικά στοιχεία για να βρούμε περισσότερες λύσεις. Ήδη αναφέρθηκα στους κατασκευαστές. Οι κανόνες ασφαλείας και εξαγωγής των ρυθμιστικών μας πλαισίων διεθνώς είναι και αυτό πολύ σημαντικό στοιχείο η επιτάχυνση της ε, διαδικασίας και των κύκλων καινοτομία και η πρόσβαση στις αγορές που μέχρι στιγμής υπήρξαν κλειστές για τις ε, επιχειρήσεις μας. Για τους αερολιμένες θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια συνολική συμφωνία με άλλες χώρες και περιφέρειες μέσω της ε, ε, αναθεώρησης ε, του κανονισμού, αλλά θα πρέπει όμως οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έχουν μια παγκόσμια, μια διεθνή προσέγγιση και στις επενδύσεις τους, ώστε να είναι παρούσες στις διεθνείς αγορές. Συμπερασματικά λοιπόν, έχει γίνει πολλή δουλειά σε αυτό τον πρώτο χρόνο, αλλά ήταν το πρώτο βήμα. Η δουλειά είναι μπροστά μας. Ελπίζω πραγματικά λοιπόν να έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο και να υπάρξετε τόσο δραστήριοι όσο υπήρξατε και κατά τη διάρκεια αυτής εδώ της πρώτης χρονιάς ώστε η ευρωπαϊκή αεροπλοεία να είναι όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική στην εσωτερική μας αγορά αλλά και διεθνώς. Και θα ήθελα να σας προσκαλέσω όλους να ελέγχετε την ιστοσελίδα γιατί όλα αυτά έχουν κωδικοποιηθεί ηλεκτρονικά και θα ήθελα να μας παρακολουθείτε, να βοηθάτε την ε, στρατηγική αυτή, διατηρώντας βεβαίως μια επικοδομητική κριτική προσέγγιση. Σας ευχαριστώ. Yeah. Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, κύριε Βιολέτα Μπούρ. Σας ακούσουμε τώρα τους συντονιστές. Ο κύριος Φαντενκάμπ έχει το λόγο πρώτος και θα δώσουμε τρία λεπτά στον καθέναν, γιατί δεν έχουμε περιοριστό χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και ήθελα ξεκινώντας να σημειώσω ότι οφείλουμε να συγχαρούμε την Επίτροπο Μπούρτς. Τη συγχαίρω λοιπόν εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος γιατί σήμερα μπορείς να μας παρουσιάσει αυτή τη δέσμη για, την, ε, ε, για τις αερομεταφορές. Μια δέσμη μέτρων περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό. Πολλά υπόθηκαν για τη δέσμη μέτρων. Πολλά θέματα έχουν ήδη συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα δούμε κατά τη διάρκεια των προσεχών μηνών εάν είναι στο, αν έρονται στο των περιστάσεων τα μέτρα αυτά. Και έτσι θα ήθελα να πω ότι μπορούμε να δούμε μια στρατηγική για τις ενέργειες μεταφορές. μια στρατηγική η οποία ξεπερνάει τον ανταγωνισμό απλώς και μόνο. Ίσως θα πρέπει να εστιαστούμε, είχα σκεφτεί εγώ αρχικά, τις ε, χώρες του Περσικού, αλλά το θέμα ξεπερνάει αυτό το ε, επίπεδο στο, στα μία επανδρομένα τελικά ε, αεροπλάνα. Οι Αμερικανοί δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη την επεξεργασία της νομοθεσίας τους. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε και το ε, σύστημα SHIFT, και την διαλειτουργική διάσταση των μεταφορών, συνδυασμό με του σιδηροδρόμου σε παραδείγματα. Και πρέπει να κοιτάξουμε και τις, μεταφορ... και τις μετακινήσεις, τα περιφερειακά αεροδρόμια, την κατανομή των πτήσεων, ε, τον υπερβολικό φόρτο πτήσεων, και βέβαια στις διμερείς συμφωνίες τη διάσταση της αμοιβαιότητας που έχει τεράστια σημασία. Υπάρχουν πολλές ε, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες που απειλούνται από τις αεροπορικές των χωρών του Περσικού. Πρέπει λοιπόν να τακτοποιήσουμε το τουίκο μας. Γι' αυτό και το θέμα των κοινωνικών σχέσεων, των εργασιακών σχέσεων έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα στη, στη σχέσει ανταγωνισμού, αλλά δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε αυτό, όπως δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και τη διάσταση του περιβάλλοντος, που έχει μεγάλη επικαιρότητα λόγω και της COP21 για τις ενέργειες ε, μη στρατιωτικές μεταφορές, για την πολιτική αεροπορία, δηλαδή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως είπε και η Επίτροπος, να ενθαρρύνουμε τον τομέα και να μην τον αποδυναμώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις να αντιμετωπίσετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά αυτή και θέλω να σας ρωτήσω το εξή. Θα περάσω κατευθείαν στα πιο επίκαιρα ζητήματα, ελπίζω ώστε να δώσω απαντήσεις. Στη σελίδα 10 στο 2, 4 σημείο, μιλάτε για την ενίσχυση του κοινωνικού θεματολογίου και τη δημιουργία ανταγωνιστικής αεροπορίας, αερομεταφορών, περιβάλλων, εργασιακές σχέσεις, απασχόληση, εργατικό δίκαιο κ.ο.κ. Ερωτώ λοιπόν τα Θα διευκρινίσει η Επιτροπή στις προτάσεις ε, ότι θα πρέπει να ισχύουν για το πλήρωμα οι συνθήκες απασχόλησης που προβλέπονται από το εγχώριο δηλαδή το δίκαιο της έδρας της αεροπορικής εταιρεία και δεύτερον και προς την ίδια κατεύθυνση διαπιστώνουμε ότι η Γενική Διεύθυνση MOVE μεταφορών έχει περιορισμένες αρμοδιότητες στον τομέα των εργασιακών σχέσεων στα κοινωνικά ζητήματα δηλαδή και ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει και η συμπεριφορά, η στάση της Γενικής Διευθύνσης για την απασχόληση υπό την Επίτροπο με το ε, πακέτο μέτρων για την κοινοτικότητα του εργατικού δυναμικού πρόσφατα, που έχει πολύ μεγάλη ε, σημασία για μας. Υποχρώθηκε λοιπόν να αποσύρει η Γενική Διεύθυνση για την απασχόληση της σχετικές προτάσεις. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχει κάποιο συσχετισμό με τα θέματα των μεταφορών. Και τρίτη ερώτηση για τον ανταγωνισμό. της προτάσης της σελίδα 4 της ανακοίνωσής σας όπου κάνετε λόγο για ε, την επεξεργασία, η επανεπεξεργασία της οδηγίας 868 το 2004. Τι θα κάνατε σε σχέση με τις διατάξεις οι οποίες ποτέ δεν υλοποιήθηκαν από ορισμένα κράτη-μέλη, γιατί ως Επιτροπή στα θεματοφύλακα των συνθήκων. Και ερωτώ επίσης ταυτόχρονα, κράτη τα οποία καλύπτουν ε, ε, μέγα ή το μείζον τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού να προβείτε σε κάποιες ειδικέ συμφωνίες για τις ενέργειες μεταφορές πώς θα ε, συμβιβαστούν όλα αυτά. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλο αίτημα να μην πληγεί η ενέργεια βιομηχανίας μας, ο ενέργειος κλάδος, ε, σε σχέση με αυτές τις προοπτικές. Ποια είναι η δική σας θέση, κυρία Επίτροπε, και μια τελευταία παρατήρηση για τη σελίδα 8, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ομιλεί για την αναγκαιότητα για επανεπεξεργασία της νομοθεσίας σε σχέση με τις υπηρεσίες εδάφου το handling. Ξέρετε ότι υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την προηγούμενη μας ε, βουλευτική περίοδο σε σχέση με την υπερνεοφιλελεύθερη προσέγγιση που είχε υιοθετηθεί. Θα κάνετε κάτι καινούριο ή θα επιμείνετε στις ε, ήδη ε, ληφθείς αποφάσεις. Ευχαριστώ Κύριε Φώστερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που σας βλέπω εδώ. Είναι όντως ευρύτατο το πακέτο αυτών μέτρων. Πρέπει να ζυγίζει και 7-8 ε, κιλά φαντάζομαι. δεν έχω μπορέσει να το δώσω όλες τις λεπτομέρειες, αλλά η επισκόπηση με το πιο σύντομο έγγραφο που μας καταθέσατε είναι αρκετά ε, διεξοδική από ό,τι βλέπω. Έχω μια-δύο παρατηρήσεις. Γιατί, όπως λέτε, έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας. Σημειώνω λοιπόν ότι ναι, θέλουμε μια κάποια κινητικότητα στη Συμφωνία για τι Ενέργειε Μεταφορέ και την υποστηρίζουμε. Πολλά από τα θέματα τα οποία εκθέσατε πιστεύω ότι αξίζει να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο και για να το συνδέσω η ιδιοκτησία και ο έλεγχο, Ξέρετε, έχει περάσει πολλή χρόνο από την εποχή που μιλήσαμε για ανοιχτού εφαίρε μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωση και ακόμα στο θέμα τη ιδιοκτησία και του ελέγχου δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά, άρα δεν μπορώ να πω ότι περιμένω συνταρακτικέ εξελίξει. Θα ήθελα όμω να το κοιτάξουμε και κυρίω προερχόμενοι από χώρα που υποστηρίζει τι ελεύθερε συναλλαγέ, δεν θα ήθελα να υπάρχουν περιορισμοί ω προ την ιδιοκτησία, γιατί κάπω έτσι τελευταία λειτουργούν οι επιχειρηματικέ δραστηριότητε και δυνατό συμβαίνει κάτι εκεί πίσω, τι γίνεται. Ε, και κάπω έτσι λειτουργούν και οι επιχειρηματικέ δραστηριότητε. Για τα σλότ βεβαίω μιλήσατε, για τι χρονοθυρίδε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά κάθε ε, βούληση που θα μπορούσε να έχει κανείς και ξέρετε ότι εγώ υποστήριζα τους ανοιχτούς εφαίρες γιατί είχα και την σχετική εισήγηση και είχα προσπαθήσει να δώσω το λεκτήριο λάκτισμα διαρωτώ με πώς μπορούμε να πιέσουμε τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να αναπτύξουν περισσότερο το δυναμικό είναι όλα πάρα πολύ καλά όταν θέλουμε να ανοίξουμε τις ενέργειες μεταφορές ε, τους ε, αεροδιαδρόμους ή πώς αλλιώς τους λέμε τα φάπια όλα αυτά το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν υπάρχει αρκετό δυναμικό επί του εδάφους Άρα λοιπόν, ό,τι και να κάνουμε, πάλι θα, βρισκόμαστε στην ίδια θέση. Το είδαμε και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε πολλά άλλα κράτη-μέλη. Για την ε, αναθεώρηση του κανονισμού τη ΙΑΤΑ, βεβαίω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και το θέμα των ε, μη επανδρομένων τηλεκατευθυνόμενων ε, αεροπλάνων. Αλλά για να διευκρινίσουμε, στην εποχή του, ε, της 11 Σεπτεμβρίου, της μέρης του 11 Σεπτεμβρίου δεν είχε ακόμα θεσπιστεί η, η η Διεθνής Ένωση για την ε, Ασφάλεια των Αερομεταφορών. Τι έχετε λοιπόν να πείτε γι' αυτό και τους όρους της ασφαλείας που έχουν να κάνουν με, τη δική σας, ε, με το δικό σας το πεδίο των Ορμοδιοτήτων ως Ευρωπαίας Επιτρόπου. Ο ανταγωνισμό. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο θέμα του ανταγωνισμού. Τι εννοείτε ω αθέμητε πρακτικέ εσεί, πώ το ορίζετε αυτό, Γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ αεροπορικέ εταιρείε με πολύ διαφορετικέ συνθήκε χρηματοδότηση ε, στον κόσμο. Και θα ήθελα να δω πώ το ορίζετε αυτό, γιατί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το πώ θα χειριστούμε τέτοια είδου θέματα. Καλό θα είναι να είμαστε προσεκτικοί στο πώ θα αντιμετωπίσουμε την ε, κατάσταση. Πρώτη πρώτα να δούμε μεγάλη προσοχή την πραγματικότητα, ώστε να μην ε, υπονομεύσουμε τι δικέ μα εταιρείε. Για το DGA, που είναι το 70% των εμπορικών ε, κινήσεων, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να το δούμε, αφορά το φορτίο και θα ήθελα και σε αυτό κάποια σχόλια από πλευρά σας. Πέραν αυτού, εκ μέρου τη ομάδα μου, των στηρητικών μεταρρυθμιστών, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την κατάθεση των προτάσεων και την έλευση σας εδώ και τόσο γρήγορα στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε και εκ μέρου των φιλελευθέρων ευχαριστούμε που ήρθατε και πριν να δείτε το Συμβούλιο. Το εκτιμούμε ιδιαίτερος όπω ξέρετε. Περιμέναμε εδώ και καιρό αυτό το πακέτο. Είπατε κι εσεί ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό ανάπτυξη για τι ενέργειε μεταφορέ, αλλά όχι απαραίτητα μέσα στην Ευρώπη. Και αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση για μα. Δηλαδή το να δούμε πώς μπορούμε να κρατήσουμε τους ρυθμούς ε, και τις εξελίξεις, ε, να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις ε, σε άλλες χώρες του κόσμου και κυρίως στις χώρες του Περσικού. Πρέπει να δούμε λοιπόν τις συνθήκες του ανταγωνισμού και κυρίως τη στρέβλωση του ανταγωνισμού που μπορεί να συμβαίνει ανά τον κόσμο. Και γι' αυτό ερωτώ πιο συγκεκριμένα Πώς νομίζετε ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια συμφωνία ή ε, διαπραγμάτευση κάποιων προτάσεων με τις χώρες του Περσικού, με την Κίνα και ούτω καθεξής. Τι είδους προτάσεις μπορείτε να καταθέσετε και πότε. Μιλήσατε για την οδηγία έγινε μάλλον λόγος για την οδηγία 868 του 2004. Πότε θα αρχίσει αυτή η αναθεώρηση, είπατε κάτι για το επόμενο έτος, αλλά το επόμενο έτος Φαντάζομαι ότι θα εννοείται την Άνοιξη, αλλά μπορεί να είναι και κάποια άλλη στιγμή. Είναι μεγάλη η χρονική περίοδο. Θα ήθελα λοιπόν να δω πιο συγκεκριμένα και είναι πολύ ενδιαφέρον για την 868, γιατί στο έγγραφό σα κάνετε λόγο για όλη την, όλο τον κλάδο των αέριων μεταφορών. Φαντάζομαι ότι οι αεροπορικέ εταιρείε έχουν τελείω διαφορετική εικόνα για την κατάσταση και για τι ανάγκε του σε σχέση με του φορεί διαχείριση αερολιμένων ή την κατασκευαστική ε, βιομηχανία. Καλό θα ήταν λοιπόν για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε ως Ευρώπη τον ανταγωνισμό μας σε όλους τους τομείς να προχωρήσουμε προς σωστή κατεύθυνση. Για τους ενιαίους ε, ευρωπαϊκούς εθέρες ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το υποστηρίζουμε και εμείς, ακόμα και από την Επιτροπή θέλουμε να το υποστηρίξουμε, αλλά θα ήταν καλό να λύσουμε και το θέμα του Γιβραλτάρ. Έχετε κάποια μυστική συνταγή ενδεχομένως. Σα έχω ξανακούσει να το λέτε. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται να απασχολεί και του Ολλανδού ω προσεχή προεδρία. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να αφήσουμε σε εκκρεμότητα. Γιατί έχει να κάνει βεβαίω ε, και με άλλα συναφή ζητήματα, όπω είναι αυτά των δικαιωμάτων των ε, επιβατών, όπω είναι τα θέματα των χρονοθυρίδων, των σλότ. Με την ΙΚΑΟ επίση θα πρέπει να δούμε πώ θα ε, αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει και την ανταγωνιστικότητά μα, πώ θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μα και ίσω θα πρέπει η Ευρώπη να ε, κοιτάξει να πάρει την πρωτοκαθεδρία στη χρήση εναλλακτικών ε, καυσίμων ε, για την προστασία του περιβάλλοντος. Για τα κοινωνικά ζητήματα και τις εργατικές θέσεις βεβαίως έχουν πολύ μεγάλη σημασία για μένα, όμως πάνω απ' όλα η ασφάλεια και η αποφυγή διακινδύνευσης έχουν την ύψιστη σημασία και πρέπει να βρούμε λύσεις γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλα αεροσκάφη μεγάλων αποστάσεων που διαθέτουν εξοπλισμό σχεδόν αυτόνομο από τον έλεγχο των υπηρεσιών που βρίσκονται στο έδαφος. Ωστόσο, τα μικρότερα αεροσκάφη δεν έχουν αντίστοιχο εξοπλισμό και έτσι δεν είναι και εύκολο να αποφύγουν τα μη ε, επανδρομένα τηλεκατευθυνόμενα οχήματα. Πώς θα μπορούσαμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά, η κυρία Μαντέλη έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα, κυρία Επίτροπε, να σας συγχαρώ, γιατί στην COP21 υπήρχε μία ημέρα αφιερωμένη ειδικά στις μεταφορές και πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή η παρέμβασή σας, όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτής δεν συζητήσαμε το θέμα των εναερίων μεταφορών που είναι πραγματικά πολύ άσχημο. Είμαστε σε COP21 και δεν συζητήθηκαν καθόλου οι αεροπορικέ μεταφορέ. Γιατί, γιατί σήμερα ο, αεροπορικό τομέα, όταν βλέπει κανεί εκπομπέ αερίων, είναι ο, αυτός που ρηπαίνει περισσότερο και αυξάνεται μάλιστα πολύ πιο ραγδαία από ό,τι τα άλλα μέσα μεταφοράς και ε, απαλλάσσεται από οποιαδήποτε μέτρα υπάρχουν για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και για την ε, προστασία του περιβάλλοντος. Ε, πραγματικά πρόκειται για αθέμητο ανταγωνισμό σε σχέση με, τους, με τις υπόλοιπες μεταφορές. Κυρία Μπούλτς, μιλήσατε για τεχνολογική πρόοδο. Κάθε τεχνολογική πρόοδος ε, δεν θα ρυθμίσει το πρόβλημα του κλίματος. Δεν ισχύει για ο κάθε τεχνολογικό, τεχνολογική πρόοδο αυτό δεν καταφέρατε να συμμετέχει ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών στο σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων. Θα το καταφέρουμε με αυτήν την πτυχή που μας προτείνεται σήμερα. Για ποιο λόγο να μην υπάρξει μια πραγματική εφαρμογή μιας, ενός φόρου κυροζήνης. Ε, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής ε, ε, τα ορυκτά καύσιμα ε, φορολογούνται, ενώ το, ε, τμήμα των, το τμήμα των αεροπορικών μεταφορών ε, μολύνει κατά 3% παραπάνω. Λοιπόν, ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θέσει επιτάπητο στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου όλα αυτά τα αριθμητικά στοιχεία, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να επηρεάσουμε το μέλλον. Κάτι ακόμη, το είπατε κι εσείς, το μεγάλο δράμα είναι η γενίκευση του κοινωνικού dumping στον ε, αεροπορικό τομέα και είναι πραγματικά εκθετική η αύξηση αυτού του ε, μέσου μεταφοράς. Ε, είναι αθέμητος ο ανταγωνισμός στο μισθολογικό κόστος, στην ανάπτυξη, όπως επίσης και των εταιριών χαμηλού κόστους, που πραγματικά είναι αποτέλεσμα ε, κρατικής υποστήριξης και κρατικών επιδοτήσεων ε, πρέπει λοιπόν να υπάρξουν σήμερα πάρα πολύ σοβαροί και αυστηροί κανόνες ε, για την ασφάλεια, το είπατε κι εσείς, ε, και για την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και για να υπάρχει και θεμητός ανταγωνισμός μεταξύ των αεροπορικών μεταφορών και για την ώρα δεν υφίσταται κάτι τέτοιο και πρέπει οπωσδήποτε να το επεξεργαστούμε κι αυτό. Και θα ολοκληρώσω, ελπίζω να μην υπερβώ πολύ το χρόνο μου, θα ήθελα κυρία Επίτροπη να με ενημερώσετε για το χρονοδιάγραμμα. Έχετε στο μυαλό σας ένα χρονοδιάγραμμα για την ε, έγκριση του πακέτου αυτού του αεροπορικού, γιατί μιλήσαμε για την τεχνολογία των drones, των μη επανδρομένων ε, ε, αεροσκαφών. Μήπως μπορείτε να μας πείτε ένα χρονοδιάγραμμα, παρακαλώ. Ο κύριος Πέτερ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να αφήξω τα πιο σημαντικά από τα στοιχεία που ακούσαμε. Για τα κοινωνικά ζητήματα είναι, νομίζω, πραγματικά είναι από τα πιο σημαντικά. Γιατί εδώ επιτρέπουμε σε πιλότους τρίτων χωρών να χρησιμοποιούν ευρωπαϊκούς αερολιμένες χωρίς να σέβονται το CSR που έχει εγκαταστήσει η ΆΣΑ. Αυτό λαμβανωμένου υπόψη και του κοινωνικού dumping που λαμβάνει η χώρα είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα Πρόβλημα το οποίο έχουμε ήδη σημειώσει πολλές φορές ή στον πλαίσιο των μεταφορών. Υπάρχουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις ε, στις ε, μεταφορές τις οδικές που έχουμε σημειώσει πολλές φορές και αυτά συμβαίνουν και στην αεροπλοεία. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε πληρέστερα και πιο αποτελεσματικά τις κοινωνικές στοχές του τομέα αυτού και αυτό για το προστατεύοντας και το μέλλον του ίδιου τομέα. Επομένω, η ερώτηση μου είναι γιατί να μην έχουν γίνει τα ίδια ε, εν είδη προστασίας όπως έχουν γίνει και για άλλους τομείς. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Επίτροπο για να απαντήσει και μετά θα έχουμε ένα δεύτερο γύρο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα ευρύτατο φάσμα ερωτήσεων. και αν ξεχάσω κάποια ερώτηση παρακαλώ να μου το θυμίσετε. Γιατί δεν έχω καμία πρόθεση να παρακάμψω καμία από τις ερωτήσεις. Λοιπόν, είπατε για κοινωνικά, ισότιμο ανταγωνισμό, περιβάλλον και γενικότερα θέματα αεροπλοείας, όπως τα ομοδοποίησα. Δύο πιο σύντομε απαντήσεις. Μια γενική για την αεροπλοεία και για τον Γιβραλτάρ πιο συγκεκριμένα. Επί του τελευταίου θα πω ότι σε αυτό είμαστε μαζί. Τα κράτη-μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν. Μέσω ενός επικοδομητικού διαλόγου και παρουσιάζοντας τις ζημίες που έχουμε με σαφή τρόπο θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση, πιστεύω. Ε, καταβάλλονται ήδη ειλικρινείς προσπάθειες και πραγματικά νομίζω ότι όλοι θα συμμετάσχουν ενεργά και θα βοηθήσουν. Γιατί μιλούμε για δισεκατομμύρια ευρώ, το έχουμε ξαναπεί, αλλά αξίζει να το επαναλαμβάνομαι και για ε, πολλές, πάρα πολλές θέσεις απασχόλησης. Και γι' αυτό ζητώ τη στήριξη όλων σας για να βρούμε μια λύση. Είναι ένα θέμα ε, κυριαρχίας, θα πρέπει να στηρίξουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά επαναλαμβάνω, οι απώλειες, οι ζημίες είναι τεράστιες. Τώρα για τα θέματα γενικής αεροπλογίας. Ναι, έχουμε συζητήσει με τους ενδιαφερόμενους φορείς και έχουμε μια σειρά από θετικά στοιχεία. Το θέμα των μη επανδρομένων τηλεκατευθυντών, των drones, σε είναι ένα από τα θέματα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αναδύονται νέα προϊόντα μέσω νέων τεχνολογιών. Από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μεταξύ άλλων. Και διατηρώντας ένα πνεύμα ανταγωνισμού, ανταγωνιστικότητος. Γιατί ένας παγκόσμιος ηγέτης θα πρέπει να παρέχει τα πρότυπα και τις συνθήκες ώστε το σύνολο του οικοσυστήματος, θα έλεγα, του κλάδου να λειτουργεί σωστά. Ταυτόχρονα ενθαρρύνουμε μία εξέλιξη του οικοστήματος αυτού ώστε να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε με τον πιο αποτελεσματικό δυνατό τρόπο νέες ιδέες και νέες τεχνολογίες για να χρησιμοποιήσουμε οικονομίες κλίμακος και όγκου. Και εδώ στηρίζομαι σε μια επικοδομητική συμφωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα. Αλλά ας πάω τώρα στις ερωτήσεις που επαναλήφθηκαν αρκετές φορές από τα μέλη για τα θέματα γενικώς απασχόλησης. Αναφερθήκατε στις ε, συνθήκες εργασίας και, τις, και την ασφάλεια. Εδώ είμαστε σε στενή συνεργασία με άλλους επιτρόπους, Γιούροβα και Τάισεν πάνω απ' όλα, που είναι συναρμόδιοι. Έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά, γνωρίζουμε τις δυσκολίες και τις προκλήσεις. και λαμβάνουμε υπόψη μας τον ε, πολλαπλασιασμό της ε, βάσης ανάλογα με τον τόπο στον οποίο ε, εργάζεται το κάθε πληρώμα για να υπάρξει καλύτερη σαφήνεια. Η γάμα δέλτα δικαιοσύνη έχει μάλλον αυτή τη στιγμή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές βελτίστων πρακτικών και θα δούμε και μια πιθανή αναθεώρηση του 2008 2008 Αυτά είναι τα δύο βήματα που ακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Ε, ότι βεβαίω πρέπει να είμαστε καινοτόμοι και να είμαστε ανοιχτοί στη χρησιμοποίηση νέων προτύπων επαγγελματικών. Αλλά δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε κανένα συγκεκριμένο βήμα χωρίς πλήρη διάλογο και συνεργασία με τους ενδιαφέρομενους κοινωνικούς φορείς. Για τις συνθήκες εργασίας δεν σχεδιάζουμε, δεν έχουμε την πρόθεση στον κανονισμό ασφαλείας και κοινωνικών ζητημάτων να συμπεριληφθούν είναι η αλήθεια ότι είναι πολύ πιο δύσκολο οι πολλαπλοί operators να ελεγχθούν από τους παραδοσιακούς και υπό την έννοια αυτή η πρότασή μας θα αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των φορέων που λειτουργούν ε, σε ένα πολυεθνικό αν θέλετε πλαίσιο και κλίμακα και θα έχουμε και ένα σύστημα μοιράσματος των ε, διεθνών των παγκόσμιων περιουσιακών στοιχείων της κάθε επιχείρησης. Υπάρχει κάποια έλλειψη αρμοδιότητος σχετικά με Συγκεκριμένε δεξιότητε που λείπουν από κάποια κράτη-μέλη και προσπαθούμε να πάμε σε αυτό το pooling τη εμπειρογνωσομοσύνης στα πλαίσια του Single European Sky. Εντό τη ΙΑΣΑ υπάρχει μια ομάδα εργασία που εξετάζει το θέμα αυτό και επί τη βάση των πορισμάτων της θα προχωρήσουμε. αλλά δεν, σε καμία περίπτωση δεν θα αφαιρέσουμε την ασφάλεια από την πρώτη θέση της προτεραιότητάς μας. Δεν πρόκειται να κάνουμε υποχωρήσεις σε καμία περίπτωση ως προς την ασφάλεια. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο ισχυρό ανταγωνιστικό χαρτί της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Και θα εξακολουθήσουμε να είμαστε πολύ σταθεροί πάνω σε αυτό από αυτού δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Τώρα η επόμενη ομάδα ερωτήσεων ήταν κάποια εχέγγυα ανταγωνιστικότητος και εδώ νομίζω ότι το πιο ισχυρό εργαλείο είναι αυτές οι γενικές συμφωνίες και θα ζητήσουμε εντολή κατάλληλη ώστε να μπορούμε ώστε να διαπραγματευόμαστε αυτές τις ε, καθολικές συμφωνίες συμβάσεις επί τη βάση της αμοιβαιότητας και των ίσων κανόνων για όλους. Αλλά σε αυτές τις διμερείς συμβάσεις κυρίως θα εστιαζόμαστε στην πρόσβαση στην αγορά, δίκαιο ανταγωνισμό και για θέματα ελέγχου και ευθύνη. Αλλά πάντοτε επί τη βάση της αμοιβαιότητας. Τον 868 τον αναθεωρούμε λέει η Επίτροπος, τον κανονισμό και εκτός των όσων ανέφερα θα συμπεριλάβουμε τις επενδύσεις, τις συνθήκες ε, απασχόλησης, τη διαχείριση κυκλοφορίας και βεβαίως τις συνθήκες αναστολής, λέει η Επίτροπος. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι είμαστε οι μόνοι αγορά διεθνώς που επιτρέπει τις ξένες επενδύσεις και ήταν ο μόνος τρόπος για να προσφέρουμε πολύ συγκεκριμένα ωφέλη στους ταξιδιώτες η Ryanair, η EasyJet και όλες αυτές οι θαυμάσιες επιχειρήσεις δεν θα ήταν εδώ αν δεν είχαμε κάνει όλα αυτά και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ωφέλειες του πλαισίου στο οποίο έχουν καταφέρει να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά. Αναφερθήκατε και στη μία εφαρμογή του 868 δεν έχει χρησιμοποιηθεί και αυτή είναι η εξήγηση για του γιατί δεν είχαμε καταγγελίες ή διαμαρτυρίες αλλά πολύ νωρίς εντός του 16 είτε θα αντικατασταθεί είτε θα αναθεωρηθεί πλήρως. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Δεν μπορώ να σας δώσω ακριβή ημερομηνία, αλλά οπωσδήποτε αυτή είναι η δέσμευσή μας. Και θα πω ανοιχτά εδώ ότι δεν είμαι υπέρ της προστασίας. Η προστασία σκοτώνει την καινοτομία, σκοτώνει το πνεύμα της ανταγωνιστικότητας, αλλά παράλληλα, και δεν φοβούμαι να το πω, είμαι υπέρ του απολύτως ελεύθερου και ανοιχτού ανταγωνισμού και είμαι σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να βρούμε εκεί μια κατάλληλη ισορροπία. Και νομίζω ότι έχουμε μια πολύ σημαντική ευκαιρία προωθώντας προς την κατεύθυνση αυτή διεθνώς. Για τα θέματα ελέγχου και ευθύνηση όπως είπα. θα προτείνω το Συμβούλιο και το Συμβούλιο έχει δείξει ότι είναι ανοιχτό σε αυτό να μας δώσει μια εντολή ώστε να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε επί τη βάση της αμοιβαιότητας και των ίσων κανόνων για όλους όπως σας είπα ήδη και θα εκδώσουμε και κατευθυντήριες γραμμές της Κομισιόν για την σωστή ερμηνεία των υφισταμένων διατάξεων και κανόνων για να έχουμε ασφάλεια δικαίου και θα ελαφρύνουμε κάποιους κανόνες εντός του πλαισίου των καθολικών αυτών συμφωνιών, των comprehensive agreements, για να το πούμε και ελληνικά. COP21 τώρα, πάρα πολύ σύντομα να αναφερθώ. Εδώ είμαστε, έχουμε δουλέψει αρκετά και θα ήθελα να μείνουμε εστιασμένοι διότι έχουμε και δύο δύσκολες εντολές να διαπραγματευτούμε. Καταρχά, επίπεδα εκπομπών διοξιδίου και τα μέτρα της αγοράς επ' αυτού. Συναντήθηκα στο Παρίσι με τον πρόεδρο της ΙΚΑΟ, ο οποίος με βεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά θα χρειαστεί πολλή δουλειά. Δεν είναι εύκολο Έχουμε διάφορα πρότυπα που αναδύονται σε ε, παγκόσμια κλίμακα. Είμαστε πεπισμένοι ότι τα μέτρα της αγοράς είναι η καλύτερη λύση. Το Φεβρουάριο θα πάω στο Μόντρεαλ όπου θα εξακολουθήσουμε να ασκούμε επιρροή και να συνεργαζόμαστε ώστε να επιτύχουμε μια θετική ελπίζω και πιστεύω συμφωνία όπου το φθινόπωρο αργά το 2016 θα υπάρξει μία σύνοδο στο Μοντρεάλ από αυτού. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι. Δεν νομίζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν αυτό ο πρώτο γύρο των ερωταποκρίσεων. Παίρνουμε και στον επόμενο, αλλά μια και μα πιέζει ο χρόνο. Και έχουμε τώρα 13 που έχουν ζητήσει να λάβουν το λόγο. Θα δώσω από ένα λεπτό για πολύ συγκεκριμένε ερωτήσει ώστε να προλάβουμε και τι απαντήσει. λόγω κάποιου προβλήματος ασθενεία σήμερα δεν έχουμε ρουμανική καμπίνα. Μπορείτε όμως να μιλήσετε ρουμανικά, δεν θα μπορείτε να τα ακούσετε. Πασκάλ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο. Καθότι δεν έχουμε χρόνο, δεν μας δώσανε, δεν μας έδωσε αρκετό χρόνο ο Πρόεδρος, να συντομεύσω. Σας ευχαριστώ για την ε, αναφορά σας στο Γιβραλτάρ. Είναι θέμα κυριαρχίας και μακάρι ο διάλογος να είναι επικοδομητικός. Τώρα έχουμε μια τελευταία απικία στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε εδώ να διευκολύνουμε λαθρεμπόριο καπνού και άλλα λαθρεμπόρια που λαμβάνουν χώρα. Εν πάση ε, δεύτερο, να περάσω στο θέμα της ασφάλειας. Έχω ασχοληθεί με αυτό όπως και άλλοι συναδελφοί, αλλά με ανησυχεί ιδιαίτερος και ανησυχεί πολύ κόσμο. Και στο, στο ψήφισμα αυτό αποτυπώθηκε και στην πρωτοβουλία μάλιστα που είχα την τιμή να ηγηθώ. Έχουμε τα θέματα των σκάνερ ασφαλείας, των υπευθύνων, των χειρισμών αυτών. Όλα αυτά τώρα είναι υπό τη σκιά των απειλών τρομοκρατικών χτυπημάτων. Και έχουμε και το PNR που είναι ε, μια ιστορική ευκαιρία θα έλεγα. Αλλά θα ευχαριστούσα την Επίτροπο που το κατέστησε αυτό, το υπογράμμισε ότι είναι από τα σαφέστερα ζητήματα. Η γενικότερη ανησυχία και το πόσο ευαίσθητος είναι ο τομέας αυτός για την προάσπιση των ελευθεριών μας. Σας ευχαριστώ. Η Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε, για την παρουσίασή σας. Ευπρόσδεκτη αυτή η στρατηγική για τις ανάγκες μεταφορές. Την περιμέναμε εδώ και καιρό. Και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εστιαστώ στις συμφωνίες με τρίτες χώρες τις τελευταίες ε, χρονιές βλέπουμε όλο και πιο σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ άλλων στην ασιατική και κινέζικη αγορά. Χρειάζεται να ε, βελτιωθεί η πρόσβασή μας στις κινέζικες αγορές. Γιατί όλο και πιο πολλοί διεθνείς φορείς έχουν δραστηριοποίηση στον τομέα των μεταφορών στην Κίνα. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι βεβαίως οι νέες τεχνολογίες, τα μη επανατρωμένα τηλεκατευθυνόμενα οχήματα και βέβαια και η συνδεσιμότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και έναντι τρίτων κρατών γιατί υπάρχουν περιοχές, πόλεις με μεγάλο δυναμικό, οικονομικό και τουριστικό που δεν έχουν ακόμη επαρκείς διασυνδέσεις. Χρειάζεται λοιπόν αυτό για να εξασφαλιστεί η πρόοδος στον τομέα αυτών στις περιοχές αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πάβελ Τελίτσκα. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Ε, είδα το πρόσωπό σας ότι ήσασταν πολύ ευχαριστημένοι και ενθουσιασμένοι θα έλεγα μάλιστα και εμείς το ίδιο για τη διαδικασία που μας, περιγράψετε, που μας περιγράψατε, κάτι το οποίο εκτίμησα ιδιαίτερα στην πρότασή σας αλλά και στην παρουσίασή σας, είναι ότι ε, είναι προσανατολισμένη περισσότερο στην ανάπτυξη, στην καινοτομία και στις επενδύσεις. Αν καταφέρουμε να προωθήσουμε αυτά τα στοιχεία, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε και τις δευτερεύουσες προτεραιότητές μας να τις επιτύχουμε. Ε, εκτιμώ επίσης το γεγονός ότι προσπαθείτε να το διασυνδέσετε και με άλλες στρατηγικές και με άλλους τομείς. Νομίζω ότι αυτό λειτουργεί πολύ καλά Τις εξής ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω. Όλες οι ερωτήσεις που αφορούσαν τον 868, την 868 με βρίσκουν σύμφωνο, αλλά το θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ε, το θέμα του πακέτου των αεροπορικών μεταφορών έχει άμεση σχέση με την οδηγία 868. Δύο σχόλια λοιπόν που θα ήθελα να κάνω είναι τα εξής. Πρώτον, αναφερθήκατε στην καινοτομία. Και αυτό συνδέεται βέβαια και με τη σχέση με άλλους τομείς και άλλες στρατηγικές και θα ήθελα να τονίσω ένα βασικό σημείο, το Γαλιλαίο. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, γιατί δεν έχω χρόνο, αλλά και απόψε ασφάλειας υπάρχει μία άμεση σχέση και δεν μιλάω για μια νέα στρατηγική για το Γαλιλαίο, γιατί το άκουσα και αυτό. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι πώς θα μπορέσουμε να παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες ε, χωρίς τη σύνδεση με τον Γαλιλαίο. Και δεύτερη ερώτηση, διαμαρτύρεται ο Πρόεδρος, ε, θα ήθελα να ρωτήσω για τη σχέση με τα μικρότερα αεροδρόμια. Ευχαριστώ, Ντανιέλα Ευχαριστώ να ευχαριστήσω και την Επίτροπο την οποία άκουσα με προσοχή. Τώρα μόλις έχω το χρόνο τον επαρκή να μελετήσω πληρέστερα το έγγραφο προγραμματισμού θα, είμαι, θα μπορέσω να είμαι πιο συγκεκριμένη αλλά σημείωσα κάποια από αυτά που λέγατε και προκύπτει μια, μια σημαντική απορία που έχω για την αρχή της αμοιβαιότητας. Εδώ έχουμε κάποιες αμφισημίες μου φαίνεται. Ε, πώς, τι, τι πρόθεση έχει εδώ η Κομισιόν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε την ε, πρώην εθνική μας, εθνικό μας μεταφορέα, που έχει γίνει πλέον ε, ιδιοκτησία σε σημαντικό ποσοστό της Etihad. Τώρα γνωρίζουμε την θέση της Κομισιόν για τις κρατικές ενισχύσεις και σωστή είναι η γενική κατεύθυνση, αλλά πώς τοποθετούμαστε όταν Συγκεκριμένε επιχειρήσεις που έχουν, που δέχονται κρατικές ενισχύσεις, προχωρούν σε αγορές άλλων επιχειρήσεων. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί δηλαδή μια στρατηγική εντός της οποίας θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ή να περιοριστεί λίγο αυτή η κατάσταση. Όχι λέει ο πρόεδρο, διακόπτη. Η Etihad είναι ολόκληρο πρόβλημα να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ. Ο Ζόρ επόμενο, χωρί μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Επίτροπε, για τι διευκρινήσει σα. Πιστεύω ότι συμμεριζόμαστε όλε τις προκλήσεις, να εξελίξουμε προκλήσουν και υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες που γεννά αυτή η στρατηγική. Τα πέντε σημεία τα οποία απαριθμίσατε είναι και τα σημαντικότερα, πιστεύω. Για μένα παραμένει ένα συγκεκριμένο ερώτημα έκρεμες. Μιλήσατε για τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν προσδιοριστεί ως μια σαφής νομοθετική προσέγγιση. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να ακολουθήσετε αυτή τη νομοθετική προσέγγιση όμως γιατί δεν βλέπω να είναι πολύ σαφή τα πράγματα ως προς τον κανονισμό 868, ότι δεν υλοποιείται, ως προς τα δικαιώματα των επιβατών. Βλέπουμε ότι απλώς λαμβάνει γνώση της νομολογίας της του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η Επιτροπή, το usual place of business, συνήθις τόπος απασχόλησης και όλα αυτά τα ζητήματα ε, φαίνεται να έχουν μείνει σε τέτοια εκκρεμότητα που να μην οδηγούν σε καμία λύση όπω έχει κατάσταση και χρειάζεται νέα νομοθετική προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο, και πάνω απ' όλα που τηρήσετε με τόση ακρίβεια τον ε, χρόνο σα. Τα υπάρχοντα πρότυπα δεν θα έπρεπε να αποδυναμωθούν, γιατί φοβόμαστε τον εξωτερικό ανταγωνισμό από χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ο κλάδο μα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε το γεγονό ότι έχουν εμπιστοσύνη οι επιβάτε σε αεροπορικές εταιρείες και δεν είμαι σίγουρη ότι είναι σωστή η προσέγγιση μεταξύ ισορροπίας μεταξύ κινδύνων και ανταγωνισμού όσον αφορά την ε, ε, αλλαγή του τρόπου μεταφορά στο modal shift εξακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος να χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό αεροπλάνου και τρένου και αυτό δεν αναφέρεται στην παρουσίασή σας. Επίσης μου φαίνεται ότι χάσαμε την ευκαιρία στο θέμα των κυρώσεων ε, γιατί η συνήθις ε, διατύπωση της ε, αποτροπής χρησιμοποιείται, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ευρωπαϊκής νομοθεσίας έχουμε ασχοληθεί και με διαδικασίες επί παραβάση και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το εξετάσουμε. Μεταξύ των οργανώσεων ε, που ανταποκρίθηκαν στις, δια, στις διαβουλεύσεις μαζί σας είχαν σοβαρές, σοβαρούς ενδιασμούς σε σχέση με την εποπτεία και αυτό δείχνει ε, άλλωστε και ε, η δική σας ε, απάντηση στη διαβούλευση. Μόνο πέντε ανάδοχοι απάντησαν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρουσίασή σας, Επίτροπε. Ε, πολλές, πολλές απόψεις ακούστηκαν σε σχέση με τα νέα μέτρα για, για τον αθέμητο ανταγωνισμό. Είναι κάτι το οποίο είπατε ότι θα το συμπεριλάβετε σε ανακοίνωση το 2016. Αν δεν κανείς την υποσημείωση 17, ανησυχώ λιγάκι, γιατί πολλές ε, χώρες πιστεύουν ότι ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Λέει ας πούμε εδώ ότι οι νομοθετικές προτάσεις θα ε, υπόκειται στην Στι στις απαιτήσεις της χρηστής διακυβέρνησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζω ότι η 868 δεν θα είναι μια υποσημείωση την οποία θα μπλοκάρει ο κύριος Τίμερμαν. Πώς μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό γιατί είναι απολύτως απαραίτητο. Δεύτερο ερώτημα, βλέποντας το έγγραφο εργασία σας που συνοδεύει την ανακοίνωση, ε, οι οι ζώνες συγκρούσεων αναφέρονται μόνο μία φορά είναι ένα θέμα το οποίο έχει άμεση, άμεση σχέση με την ασφάλεια και για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το εξετάζει περισσότερο και δεν το πραγματεύεται περισσότερο σε, στην ανακοίνωσή της. thank you very much, Commissioner. I'm delighted that we've come to this point, and I hope you, you have, I'm sure you have absolutely the same sense of enthusiasm that we have here, here for your, for your package. There's just um, you've lots, lots of areas. I'm interested in two particular areas. My time is short. Just on the um,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 Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ μία ερώτηση έχω να θέσω στην Επίτροπο. Στη στρατηγική την οποία αναπτύσσεται βλέπετε, βλέπω ότι ο ανταγωνισμός και ο αθέμητος ανταγωνισμός είναι σημαντικό σημείο. Το θέμα των καυσίμων θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτον, το πρώτο θέμα που ήδη ετέθη, το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή θεωρείται επαρκές, θα τροποποιηθεί ή θα είναι το αντικείμενο μιας νέας ε, πρότασης για το σύνολο αυτών των συμφωνιών. Δεύτερον, επειδή αυτές οι συμφωνίες για ε, ε, πραγμάτευσή τους γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχετε ως προτεραιότητα, έχετε προτεραιότητα συγκεκριμένη για αυτές τις συμφωνίες, από πού ξεκινάμε. Επίσης, θα μας δώσετε προθεσμίες για να γνωρίζουμε πόσο χρόνο θα, γίνονται, θα πάρουν οι διαπραγματεύσεις και ποιο είναι το αντικείμενο. Και επίσης, αν έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία για να υπάρξουν τόσες πολλές διαπραγματεύσεις παρα, ε, παράλληλα, γιατί για μερικές χώρες είναι πάρα πολύ επίγον το θέμα. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την παρουσίαση. Υπάρχει το θέμα των κοινωνικών ζητημάτων, όπως είπατε κι εσείς. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές γι' αυτά. Δεν υπάρχει αρκετή ανταπόκριση όσον αφορά τα κοινωνικά ζητήματα. Οι διεθνείς συμφωνίες σημαίνουν όλο και περισσότερα πληρώματα τρίτων χωρών. Αρχίζουμε σιγά σιγά και στην Ευρώπη να έχουμε πληρώματα με βάση ε, στο ε, με βάση στον, ε, στη Δομινικανή Δημοκρατία και θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών, πώς ακριβώς ε, θα το συνδυάσουμε αυτό με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Επίσης, για τα καύσιμα, υπάρχουν καινοτόμα καύσιμα, υπάρχουν ε, ε, καινοτομίες στον τομέα των καυσίμων που τις συζητούμε σε άλλους τομείς, αλλά όχι στην αεροπορία. Υπάρχει το θέμα της κυκλικής οικονομίας. Ο κύριος Τίμερμαντ το ανέφερε αυτό στις παρουσιάσεις του. Υπάρχουν πάρα πολλά αεροσκάφη που κατά το 2016 θα είναι πλέον πάρα πολύ μεγάλα σε ηλικία και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Όσον αφορά τον κίνδυνο τώρα, θα μπορούμε να προβούμε σε έρευνες όσον αφορά τις, ε, των ατυχημάτων, όπως τη Εσπανέργεια παράδειγμα, όταν είχε συμβεί, τότε ε, τι θα κάνουμε αν οι εθνικές ερευνητικές επιτροπές ε, δεν έχουν επαρκή αποτελέσματα. Ο κύριος Νίλσεν έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ την Επίτροπο που ήρθε να μας μιλήσει. Υπάρχει μια πρόταση που θα πρέπει βέβαια να υλοποιηθεί στην πράξη. Ο διάβολος ξέρουμε ότι κρύβεται στις λεπτομέρειες και από εκεί θα κρυθούν πολλά. Ρωτώ λοιπόν, ο διάλογος, ο κοινωνικός διάλογος έχει σημασία επαρκή για εσάς, είναι σημαντικά τα εργασιακά ζητήματα θα ε, κρυθεί ως κρίσιμος ο συσχετισμός μεταξύ συνθήκων απασχόλησης και ασφάλειας των πτήσεων. Είναι νομίζω λίγα τα ζητήματα για τα οποία είναι ο κόσμος ομόφωνος. Και ένα από αυτά είναι ότι χρειαζόμαστε πιο ασφαλείς πτήσεις. Σε αυτό θα ήθελα λοιπόν να μου δώσετε απάντηση. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να διατυπώσω μια ερώτηση. Cheap flights, φθηνές πτήσεις. Ναι, μπορεί να είναι αυτό στόχο, δηλαδή για 23 ευρώ να αγοράζω ένα αεροπλάνο να, ένα <laughs> αεροπορικό ειστήριο και να ταξιδεύω από τι Βρυξέλλες για το Βερολίνο, ενώ είναι πενταπλάσιο το κόστος ενός εισιτηρίου με το τρένο. Μπορούμε αυτό να το δούμε ανεξάρτητα από το κόστος για το περιβάλλον. Και επίσης υπάρχει και ανταγωνισμός, ο ανταγωνισμός μέσα στον τομέα των εναέριων μεταφορών. Αν είχαμε κάνει μια σωστή κατανομή, θα είχαμε ε, ίσως καλύτερες συνθήκες ανταγωνισμού, γιατί η Φερρυπίν διόδια δεν... Ε, χρεώνουν τα αεροπορικά ταξίδια, εκτός από τη Σιβηρία. Στο 15-16% από την άλλη είναι η επιβάρυνση για κάθε στάση σε σταθμό των ε, τρένων. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ, έχετε ανοίξει το βλέμμα περισσότερο ώστε να μην ρυθμίσετε τον κάθε τομέα χωριστά, αλλά να κοιτάξετε το μέτρο μεταφορών σαν σύνολο και να έχουμε πιο υγιή ανταγωνισμό, πιο θεμητό ανταγωνισμό, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα νομίζω ότι έχετε τι 13 ερωτήσεις σας και περιμένουμε τις απαντήσεις με ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Πέντε λεπτά έχουμε. Και είναι πολλά τα ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν συντομότερη. Ο κύριος Μαρινέσκου θέλει να κάνει μια ερώτηση. Ναι, με ξεχάσατε κύριε Πρόεδρε. Ε, εντάξει, δεν περάζει. Λοιπόν, αναφέρατε, αναφέρετε στη, σελίδα 6, κάνετε έκκληση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για να εγκρίνει τον Ευρωπαίο ε, ενιαίο ουρανό. Ξέρετε ότι αυτό θα πρέπει να το πείτε στο Συμβούλιο, ε, εκείνοι μπλοκάρουν τις διαδικασίες. Υπάρχει μια γενική προσέγγιση και δεν άρχισαν οι διαπραγματεύσεις και δεν είδα ούτε από την Ολλανδική κυβέρνηση ε, είδα, από την Ολλανδική Προεδρία είδα να υπάρχει σκοπός να γίνει κάτι. Ε, και έχω και ένα ακόμη ερώτημα. Τι θα γίνει με την τροποποίηση του κανονισμού της ΕΑΖΑ που έχει μπλοκάρει στο Συμβούλιο γιατί τη 216 την ανακαλέσατε και αναφερθήκατε στην τροποποίηση αυτή ε, στη σελίδα 6 οπότε είπατε ότι μπορεί να αλλάξετε το όνομα ε, να επιστρέψει στην ονομασία ΕΑΖΑ Τώρα με καθησυχάσατε γιατί αναρωτιόμουν θα μιλήσει ο κύριος Μαρινέσκου. Έτσι λοιπόν, αισθάνομαι πιο ήσυχο τώρα και παρακαλώ να λάβετε το λόγο κυρία Μπούρτσου. Λοιπόν, κάποια ερωτήματα υπήρξαν επί της φορολόγησης. Εδώ είναι βεβαίω θέμα των κρατών μελών. Αλλά με τον κύριο Μοσκοβισή έχουμε συνομιλήσει αρκετές φορές για το θέμα αυτό και διερευνούμε δυνατότητες του πώς θα μπορούσαμε να επιφέρουμε κάποια τάξη τηρώντας την αναλογικότητα εδώ. Αλλά το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θα είναι μια δύσκολη συζήτηση αυτή που θα πρέπει να γίνει με τα κράτη-μέλη, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε την προσπάθεια. Τώρα, για το modality, γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται στη στρατηγική. Είναι στρατηγική επί της αεροπλοείας και είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο αυτό και ψάχνουμε ποιο χρόνο θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε στα intermodality και ποιες ε, δυνατότητες, ε, λύσεις εναλλακτικές θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε. Αλλά η προϋπόθεση είναι η ψηφιοποίηση σε όλα τα μεταφορικά μέσα. έχοντας μια ενιαία υπηρεσία. Και γνωρίζετε ότι θα έχουμε και δέσμη επί των ε, οδικών μεταφορών του χρόνου. Επομένως με την ψηφιοποίηση και των σιδηροδρόμων σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε μια οριζόντια πλατφόρμα ώστε η συντροπικότητα να είναι πολύ πιο παρούσα σε όλες τις μεταφορές γιατί πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας την οπτική του επιβάτη. Πώς μπορεί να έχει ένα ενιαίο εισιτήριο, μια ενιαία υπηρεσία και ενιαίες δομές ε, διαχείρισης της υπηρεσίας για οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς. Τώρα, Είχαμε, είχαμε κάποιες ε, θετικές ε, ενδείξεις και νομίζω ότι υπήρχε και μία συζήτηση πριν από δύο μέρες στην Κορεπέρ και η Προεδρία του Λουξεμβούργου ακόμα και αργά το έφερε το θέμα και θα είμαι η πρώτη που θα, θα δηλώσει ικανοποιημένη αν φτάσουμε σε μια ολοκλήρωση του ζητήματος αυτού για τους επιβάτες δηλαδή σε άμεσο τράνζιτ τα περιφερειακά αεροδρόμια επίσης η Ευρώπη είναι αλήθεια έχει πάρα πολλούς αερολιμένες και πολλοί από αυτούς δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς Έχουμε όμως συμφόρηση σε πολλούς υφιστάμενους αερολιμένες και ελπίζουμε ότι κάποιοι από τους περιφερειακούς μέσω αναδιανομής της κυκλοφορίας θα κερδίσουν έδαφος. Και μέσω αερομεταφορέων πιο χαμηλού κόστους εξαναβλέπουμε την κατανομή του φόρτου κυκλοφορίας στο σύνολο των αερολιμένων. Αλλά για κάποιους από αυτούς, αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε είναι να μην έχουμε, για να το πω έτσι, αεροδρόμια φαντάσματα. Αυτό δεν θα μας άρεσε καθόλου. Θα συνδυάσουμε το σύστημα με εκείνα των σιδηροδρόμων για να μπορούμε να συνδέουμε τις, ε, τα αστικά κέντρα που δεν έχουν αεροδρόμια και που δεν έχουν και επαρκείς λόγους να αναπτύξουν αεροδρόμια, ώστε να δημιουργήσουμε κομβικά σημεία μεταφορών για να συνδέονται και αυτές, αυτές οι πόλεις. Και εκεί χρειάζεται ένας μηχανισμός επενδύσεων. Η επόμενη ερώτηση είχε σχέση με τα πολυτροπικά. Χρηματοδοτικός πώς μέσω του ΣΕΦ και του ΤΕΝΤΗ διοχετεύουμε και θα έχουμε και μια νέα σύμβαση τον Ιανουάριο για την καλύτερη συνεργασία και στην καινοτομία στον τομέα της αεροπλογίας και νομίζω ότι αυτό θα είναι άλλη μια όθηση προς επενδύσεις και σε αυτό το πεδίο. Πέραν αυτού, οι αερομεταφορές ε, διατροπικός λαμβάνουν υπόψη πάνω απ' όλα το, τον, το TNT και το ΣΕΦ ως ε, χρηματοδοτικά μέσα και μηχανισμούς. Να δούμε πως ξέχασα κάτι λέει η Επίτροπος. Ναι, τα θέματα ασφαλείας. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση, το επαναλαμβάνω ακόμα μία φορά, να θέσουμε να αμφιβόλο το επίπεδο ασφαλείας μας. Έχουμε νέες προκλήσεις και είμαστε απολύτως υπέρ της προσέγγισης ε, επί τη βάση του κινδύνου και να έχουμε ενιαία θηρίδα για την ασφάλεια. Εδώ η τεχνολογία μας βοηθάει και έχουμε κάποιες ε, δοκιμές, έχουμε κάποια τεστ σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που, τα οποία μας βοηθούν να προχωρήσουμε προς τα εμπρός, κερδίζοντας εμπειρία, αλλά και βελτιώνοντας τον έλεγχο ασφαλείας. Γιατί θα πρέπει να ε, ε, εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τις καλύτερες και τις ε, βραχύτερες δυνατές συνδέσεις ελέγχων ασφαλείας. Αυτά ξέρετε ότι τα συντονίζει και ο κύριος Αβραμόπουλος στα πλαίσια της Γενικής Δέσμης για την Ασφάλεια και συνεργαζόμαστε μαζί τους για να έχουμε την καλύτερη δυνατή ισορροπία. Κρατικές ενισχύσεις. Ξέρετε ότι έχουμε κανονισμό ισχυρό και παρακολουθούμε τις κρατικές ενισχύσεις πραγματοποιεί και για τους αερολιμένες δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε ευρύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο οι φυστάμενε διατάξεις είναι επαρκής και για την υλοποίηση της στρατηγικής εγώ υπογράμμισα που θεωρούμε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ή συμπλήρωσης και από το Συμβούλιο το ξαναλέω θα τους, δώσω, θα τους ζητήσουμε να μας δώσουν επαρκή ευελιξία διαπραγμάτευσης στην εντολή για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να αναπτύξουμε τη στρατηγική εντός των ε, ορίων που την παρουσίασε. Λοιπόν, τώρα βλέπω ότι έχετε πολλή δουλειά μπροστά σας ε, και έχουμε καθυστερήσει. Ό,τι ερώτηση έχετε παρακαλώ να μου την αποστείλετε και με χαρά να σας εξηγήσω περαιτέρω τυχέ τη στρατηγική. Ευχαριστώ για την υπομονή σα. Και βεβαίω ευχαριστώ όλου αυτού που διατύπωσαν τι ερωτήσει του και έτσι έλαβαν μέρο στη συζήτηση. Ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση και κάνουμε την διακοπή για να συνεχίσουμε.